Um, Συνάδελφοι, πριν περάσουμε στο βασικό σημείο, έχουμε ορισμένες ανακοινώσεις. Έχουμε ένα βασικό θέμα, την ακρόαση για τη Ρουμανία και καλωσορίζουμε τον Φραν Τίμερμανς, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Θα ήθελα όμως να κάνω ορισμένες ανακοινώσεις. Έγκριση μερίσιας διάταξης εγκρίνεται αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ως προς το γλωσσικό υπάρχει διερμηνία από αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, ελληνικά, τσεχικά, πολωνικά και ρουμανικά. Πορτογαλικά και σουηδικά θα είναι μόνο παθητικές γλώσσες. Τώρα, ως προς τους συντονιστές. Έχουμε διορισμούς ε, εισηγητών. Η Χέλγκα Στίβεν, ορίστηκε εισηγήτρια για την πρόταση κανονισμού για την ε, ε, αναχέτηση της διάδοσης στοιχείων τρομοκρατικού περιεχομένου. Μόνικα Μακοβέη στην έκθεση, για την έκθεση πληροφοριών και τεχνολογιών σε σχέση με την Νορβηγία, Ισλανδία και Λίχτενστάιν, Πίτερ Νίντερ Μίλλερ για την πρόταση ε, για το άσυλο σε σχέση με την ε, απόφαση καταλληλότητας για την ε, Ιαπωνία. Επίσης, η πλειοψηφία των συντονιστών αποφάσισε να προετοιμάσει ένα ψήφισμα συμβαδίζοντας με τα δεδομένα της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ε, δέχεστε αυτές, ε, αυτούς τους διορισμούς των εισήγητων και την ε, τελευταία πρόταση καταλληλότητας. Λοιπόν, διόρθωση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον οργανισμό σε σχέση με την επιχειρησιακή διαχείριση των συστημάτων ευρείας κλίμακας. Πρέπει να τα διαβάσω αυτά και ας είναι βαρετά μετά από τη συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου το κείμενο εγκρίθηκε από τη ΛΥΜΠΕ και την Ολομέλεια. Συνεπώς η διόρθωση αυτή γίνεται έτσι ώστε να γίνουν γλωσσικές διορθώσεις για να υπάρξει ε, γλωσσική και ετοιμολογική συμμόρφωση του κοιμίου. Αυτό αφορά και το Ηνωμένο Βασίλειο και το γεγονός ότι η Ιρλανδία δεν λαμβάνει μέρος. Όλα αυτά εγκρίθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου και διαβιβάστηκαν. Δυνάμει του κανονισμού 23.1 υπάρχει ένα σφάλμα στο κείμενο του Κοινοβουλίου και γι' αυτό το Κοινοβούλιο θα στείλει διορθωτικό. Και ε, αυτή η διόρθωση θα ψηφιστεί δυνάμει του κανόνα 231 παράγραφος 3. Ε, θα ήθελε κανείς να ψηφίσουμε αυτό το έγγραφο. Ε, Κατάλαβε κανένα τη διάβασα, μάλλον όχι. Λοιπόν, ε, Β, φτάνουμε στο κατώτερο κατόφλι του ενός εικοστού δηλαδή τρία μέλη και θα ψηφιστεί το έγγραφο αν χρειαστεί στις 12.30. Δεν, δεν ζητήθηκε όμως άρα δεν θα ψηφιστεί. Και τώρα ως προς τις κατεξιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2018 το Κοινοβούλιο έλαβε τις εξής αποφάσεις, εκτελεστικές αποφάσεις σε σχέση με τα έγγραφα τα οποία θα υποβάλουν οι ετούντες για θεωρήσεις μικρής διάρκειας στην Βολιβία, Εκουαδόρ, Πακιστάν και Νότιο Κορέα. Αυτό αφορά και τις θεωρήσεις για, τη, ε, για την Σαουδική Αραβία και θα πρέπει να συλλέγονται στοιχεία από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να έχουμε στατιστικά στοιχεία για την ε, εισδοχή και έξοδο αυτών των στοιχείων. Ε, η γραμματεία κοινοποίησε αυτά τα στοιχεία με email. Εάν κάποιο μέλος θέλει να αναφερθεί σε αυτό και να ε, προβάλλει μία αντίρρηση, θα πρέπει να το κάνει πριν από τις 9 Οκτωβρίου στις 12. Ε, τα διάβασα όλα αυτά για να ησυχάσετε στο μεταξύ. Τώρα λοιπόν φτάνουμε στο βασικό σημείο της ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Στρασβούργο. Έχουμε τις, την ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον πρώτο αντιπρόεδρο Φρανς Τίμερμαν. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 αποφασίσαμε να καλέσουμε τον πρώτο αντιπρόεδρο Τίμερμανς για ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στη Ρουμανία, σε σχέση δηλαδή με την ανεξαρτησία του δικαστικού τομέα. Η εντολή μας αφορά το να ακούσουμε τον Επίτροπο και μετά θα έχουμε μία συζήτηση ως προς τη δική του ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση δίνω το λόγο στον πρώτο αντιπρόεδρο, τον ε, καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που δεχτήκατε την, την πρόσκλησή μας. Ευχαριστώ. Όταν συζητήσαμε το θέμα της Ρουμανίας ήταν το Φεβρουάριο. και Μιλήσαμε για την ε, νόμη τάξη και είχαμε την ε, ευκαιρία να διαπιστώσουμε τις εξελίξεις τους ε, τελευταίους μήνες. Και έχουμε όλη την εντύπωση την πρωτοβουλία που έλαβαν οι Ρουμανικές αρχές σε σχέση με τη μεταρρύθμιση των δικαστικών διαδικασιών, των ποινικό δίκαιο και οδήγησαν σε κάποιες ε, ανησυχίες εκ μέρους πολλών φορέων τόσο στο εσωτερικό της Ρουμανίας όσο και στην Ευρώπη και διεθνώς. Πολλοί Ρουμάνοι ανησυχούν ότι οι αλλαγές που προτείνονται για τους νόμους αυτούς ενδεχομένως θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες καταπολέμησης διαφθοράς και την ε, ανεξαρτησία της ε, δικαιοσύνης. Και αυτές είναι ανησυχίες τις οποίες συμμερίζεται και η Επιτροπή. Όσον αφορά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και την, το σεβασμό των θεμελιωδών αρχών, η Επιτροπή θέλει να παρέμβει στη βάση μιας προσεκτικής ανάλυσης. Εστιάσαμε την προσοχή μας σε αποτελεσματικά μέτρα και ξεκινήσαμε έναν διάλογο με τις αρχές της Ρουμανίας. Η... Ε, Αυτές γίνουν για την ε, Ρουμανία εξίσου όπως και για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Όσον αφορά τι ανησυχίε, χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα να προσεγγίσουμε προβλήματα τα οποία θεωρήσαμε ε, ότι θα πρέπει να λυθούν με τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία. Τώρα θα αναφερθώ στι σημαντικέ εξελίξει στη Ρουμανία. Καταρχήν, οι νόμοι από το 2014 σχετικά αφορά τη δικαιοσύνη που αφορούν το καθεστώς των δικαστών και οργανώνουν το δικαστικό σύστημα και το ανάπτυτο δικαστικό συμβούλιο. Ε, το τέλος του ε, περασμένου έτους ε, τροποποιήθηκαν οι αλλαγές αυτές, αλλά το συνταγματικό δικαστήριο άσκησε, έφεση, επέκρινε αυτές τις ε, αλλαγές. Ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, ενέκρινε μία έκθεση το Μάρτιο ασκώντας κριτική στη Ρουμανία και εκδόθηκε μια γνωμοδότηση τον Ιούλιο με σοβαρέ ενισχύσει όσον αφορά την εξαρτησία του δικαστικού σώματο, την αποτελεσματικότητά του και το, την ποιότητά του. Και διατύπωσε πολλέ ε, συστάσει. Η τελική γνωμοδότηση θα εγκριθεί τέλη του μήνα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα ασχοληθεί πολύ με αυτή την γνωμοδότηση, όσο και η Επιτροπή. Ε, γεγονός είναι ότι το Ρωμανικό Κοινοβούλιο μέχρι στιγμή δεν έδειξε ενδείξει ανταπόκριση προς τις γνώμες και συστάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμή. Οι δυνατότητε ε, ε, περαιτέρω προσφυγής στα δικαστήρια έχουν εξαντληθεί. Ένα από τα τρία νομοσχέδια έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Δεύτερον, όσον αφορά τον ποινικό δικονομικό κώδικα. Το Μάιο το Ρουμανικό Κοινοβούλιο ξεκίνησε μια διαδικασία αναθεώρησης αυτού του κώδικα. Πέρασαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Οι Ρουμανικές ε, Αρχές Εφαρμογής του Δικαίου καθώς και άλλες ε, χώρες εξέφρασαν ε, ανησυχίες. Όσον αφορά ε, ε, ε, τον Οκτώβριο, μέσα του Οκτωβρίου θα υπάρξουν κάποια σχόλια. Τα νομοσχέδια αυτά είναι σημαντικά όσον αφορά την δυνατότητα των εισαγγελέων να διερευνούν και των δικαστών να καταδικάζουν φαινόμενα υψηλού επίπεδου διαφθοράς ε, στηριζόμενοι στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τη δίωξη, την αποτελεσματική δίωξη του εγκλήματος Ωστόσο υπάρχουν εδώ πολλές ε, ανησυχίες γιατί προποτείται μια αμερόληπτη έρευνα. Αλλά όσον αφορά τις ε, εθνικές αρχές και το Ρωμανικό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να επιβλέπουν το έργο επίσης των υπηρεσιών πληροφοριών, κάτι το οποίο εγείρει πολλές ανησυχίες. Ε, και υπάρχει ένα αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητά τη καταπολέμηση διαφθορά. Γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή συζητά σε τακτά χρονικά διαστήματα με τη ρουμανική κυβέρνηση σε υψηλό επίπεδο και δημοσιοποιεί τι ανησυχίε τη. Εξετάσαμε το κείμενο το οποίο πέρασε το Ρουμανικό Κοινοβούλιο και σημειώσαμε τι κριτικέ που άσκησαν άλλε χώρε μέλη και άλλοι διεθνεί φορεί προκειμένου να αξιολογήσουμε πλήρου την, ε, ε, τις συνέπειές τους ε, ζητώντας διευκρινήσεις προς την ερμηνεία των εδαφείων αυτών των νόμων. Όσον αφορά την... Και επίση θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση τη της εισαγγελία. Το Φεβρουάριο ξεκίνησα μια διαδικασία Ξεκίνησε η Ρωμανία μια διαδικασία ε, απόλυσης του ανώτατο εισαγγελέα. Τώρα, την τελική απόφαση θα λάβει ο πρόεδρος της Ρεμανίας, ο οποίος ε, στην αρχή αρνήθηκε ε, να το πράξει. Το συνταγματικό δικαστήριο ωστόσο μπορεί να υποχρεώσει τον πρόεδρο να συμφωνήσει. Σαν αποτέλεσμα ο επικεφαλής της υπηρεσίας της εισαγγελία απολύθηκε τον Ιούλιο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ότι ε, ε, υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί παλήθευσης και διαδικασίες για την ε, απόλυση των ανώτατων αξιωματούχων στο δικαστικό σώμα. Οι Ρουμανικές αρχές ζήτησαν τη βοήθεια της Επιτροπής της Βενετίας στο θέμα αυτό. Και αυτό, αυτή παραμένει μια από τις συστάσεις όσον αφορά το μηχανισμό επαλήθευσης της συνεργασίας που δεν έχει εφαρμοστεί στην περίπτωση αυτή της Ρωμανίας ε, και υπάρχουν ε, πολλέ ε, ανησυχίε σε σχέση με την κατάσταση αυτή. Τέλο, όσον αφορά άλλε εξελίξει, η Επιτροπή επίση εξετάζει κατά πόσο ε, πώς ε, χρησιμοποιούνται τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρουμανία, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο οι διαδικασίε προστατεύουν αποτελεσματικά τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Αυτό αφορά τι τροποποιήσει στο ελεγκτικό συνέδριο, καθώ και του κανόνε όσον αφορά την αρεσιμότητα στην δημόσια διοίκηση. Ε, αλλαγές που θα έχουν αποτέλεσμα στην εύρυθμη λειτουργία των εθνικών υπηρεσιών που είναι υπεύθυνε για τη διαχείριση των ενωσιακών κονδυλίων θα ε, προκαλέσουν μια άμεση αντίδραση εκ μέρου τη Επιτροπής. Αξιότιμα μέλη, εν κατακλείδη, η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματο και η δυνατότητα αποτελεσματική πάταξη τη ε, διαφθορά ε, σχετίζονται με το βαθμό προόδου τη Ρουμανία στον μηχανισμό αξιολόγηση τη συνεργασία. Είδαμε κάποια πρόοδο στο παρελθόν, ορισμένε φορέ θεματικέ πρόοδου, αλλά τώρα υπάρχει ένα κίνδυνο γιατί υπάρχει μια πραγματική επιστοδρόμηση στη Ρουμανία. Και αυτό θα είναι επιζήμιο όχι μόνο για την δημοκρατία της Ρουμανίας, αλλά και για τη θέση της ε, Ρουμανίας ως χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η, Επιτροπή κάλεσε κατ' επανάληψη τις αρχές της Ρουμανίας να δημιουργήσουν μια πλατιά συνένεση εν σχέση με το πώς θα πρέπει να προχωρήσουν στο μέλλον. Θα ήθελα να υπογραμμίσω και πάλι ότι η Επιτροπή πάντοτε είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις Ρωμανικές αρχές και να τις υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή. Και αυτό ήταν το πνεύμα υπό το οποίο επισκέφθηκα το Βουκουρέστι την Άνοιξη και είχα πολλές συναντήσεις με, με την Πρωθυπουργό της Ρουμανίας και την ηγεσία των δύο κοινοβουλευτικών σωμάτων. Ωστόσο, θα πρέπει να πω ότι η πρόσφατη εξελίξεις είναι πηγή σοβαρών ανησυχιών τόσο για μας όσο και για τους διαδηλωτές τους δρόμους της Ρουμανίας και όλους μας ε, σοκάρει η αντίδραση των υπηρεσιών ασφαλείας ε, προς τους ηρωνικούς ε, διαδηλωτές και ελπίζουμε τέτοια φαινόμενα να μην επανεληφθούν. Όπως είπα προηγουμένως σε μια άλλη συζήτηση, η χρήση βίας ποτέ δεν είναι ενδεχμένη λύση στην πολιτική. Ασφαλώς όχι και σίγουρα όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται στο κράτος δικαίου. Εάν ε, εγκριθούν αυτά τα μέτρα, τα αποτελέσματα των ε, μεταρρυθμίσεων του δικαστικού σώματος ε, θα έχουν αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά στη δυνατότητα της δικαιοσύνης να πατάξει τη διαδευθορά. Και αυτό είναι τεράστια σημασία γιατί τόσα πολλά έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο του αγώνα κατά πολέμηση διαφθορά στη Ρουμανία. Αυτό θα σήμαινε ε, μια σοβαρή παρέκκληση από θετική αξιολόγηση που έκανε η Κομισιόν τον Ιανουάριο ε, του 2017. Ε, ωστόσο, οι νόμοι δεν έχουν ακόμα εκδοθεί, άρα υπάρχει ένα περιθώριο. Η Ρουμανία θα πρέπει να... Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα κείμενα των νόμων και θα δούμε και θα εκπονηθεί μια σχετική έκθεση. Ε, γιατί σίγουρα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Όλες οι εξελίξεις θα αξιολογηθούν σοβαρά και θα συμπεριληφθούν σε αυτή την έκθεση. Όπως είπαμε κατά επανάληψη, μια αποσοδρόμηση θα αποτελέσει σοβαρή πηγή, απογοήτευσης, πηγή σοβαρής απογοήτευσης για όλους τους φίλους της Ρουμανίας. Γιατί πρόοδοι έχουν μεν ε, τελεστεί, αλλά δεν είναι μη αναστρέψιμη. Οι πρόσφατες εξελίξεις υπονομεύουν το κοινό μας στόχο να υπάρξει μια βιώσιμη εξέλιξη στην ε, Ρουμανία ούτως ώστε να μην χρειάζεται ένας μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου, γιατί πραγματικά θα ήταν μια τραγωδία αν το τελευταίο χιλιόμετρο του μαραθωνίου ε, θα πάψει ο βασικός ε, δρομέας, θα διακόψει τον, ε, ε, τον αγώνα του. Εάν οι νόμοι που έχουν συμφωνηθεί στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραβιαστούν, θα προσαχθεί η κυβέρνηση της Ρουμανίας και μέρους της, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δικαστήριο. Και Συγκεκριμένα, ε, όσον αφορά την ε, σύσταση του Ιανουαρίου 2017, ε, υπάρχει ακόμα μία δυνατότητα αναστροφής της πορείας, αλλά εναπόκειται στα χέρια ε, και στην, ε, να πω και στη βούληση των ε, ρουμανικών αρχών και θεσμών. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως θα πρέπει να ξεπεράσουμε το χρόνο και τότε δεν θα έχουμε διερμηνία. Τώρα θα θέλουμε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Τίμερμανς. Έχουμε 19 συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. για την ώρα. Θα αρχίσουμε. Κύριε Τσιουρακ, είσαστε στον κατάλογο. Θα αρχίσουμε με τους ε, συντονιστές. Δεν είναι όλοι εδώ. Όλες οι πολιτικές ομάδες αντιπροσωπεύονται. Αρχίζουμε με την κυρία Μετσούλα. Είναι εδώ. Περνά, όχι. Ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό. Με συγχωρείτε που είμαι τόσο απειλητικός, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, να συγκεντρωθώ σε δύο-τρία θέματα. Το θέμα για τη διαφθορά. Χαίρομαι που είπατε ότι η Ρουμανία κατέβαλε τρομερές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχει η εντύπωση αλλάζει τώρα. Νομίζετε ότι όλοι οι νόμοι καταπολέμησης της διαφθοράς είναι πρόβλημα και θα έπρεπε να αναθεωρηθούν ή υπάρχουν μερικές θετικές εξελίξεις που μπορούμε να αναφέρουμε σχετικά με τις πληροφορίες. Θυμόμαστε το μυστικό πρωτόκολλο και οι πληροφορίες που είχαν ε, από αυτό το πρωτόκολλο και που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Πώς νομίζετε ότι μπορούν να υπάρξουν διατάξεις τώρα, υπάρχουν καλά παραδείγματα από άλλα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα για τις ε, εκδηλώσεις είχαμε στην Γερμανία παραδείγματα όπου ένας μικρός αριθμός διαδηλωτών πόρεσαν να αλλάξουν μια ειρηνική διαδήλωση σε κάτι που είναι το αντίθετο και βίαιο, οδηγώντας στην βία. υπήρξαν έρευνες και συνέπειες. Υπάρχει κάτι τέτοιο σχετικά με τις διαδηλώσεις στη Ρουμανία και η τελευταία ερώτηση, συμφωνείτε ότι ήρθε η ώρα να χρησιμοποιηθεί ο μόνιμος μηχανισμός για το κράτος δικαίου και να ε, μην ε, συγκεντρωνόμαστε μόνο σε ένα κράτος μέλο. ECR, συντονιστής. Ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. κύριε Πρόεδρε. Ναι, υπήρχαν και διαδηλώσεις ειρηνικές που εκφυλίστηκαν και κατέληξαν με βία. θέλησαν να διαδηλώσουν εναντίον των διεφθαρμένων αρχών. Ορισμένες προσπάθειες καταβλήθηκαν από δημοσιογράφους ε, για να μπορέσουν να δουν τι συμβαίνει. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί με ε, δακρυγόνα, με ε, σωλήνες, με νερά, τότε υπήρξε βία και δεν υπήρξε καμία αιτιολόγηση των πράξεων αυτών. Ένας είπε ότι η βία ήταν νόμιμη και αναγκαία. Αυτό σημαίνει ότι, ότι η Ρουμανία έχει παρεκκλίνει. Θα πρέπει να παταχθεί η διαφθορά στην Ρουμανία και θα πρέπει επίσης να ασχοληθούμε με τις υπηρεσίες πληροφοριών που εργάζονται με τρόπο που δεν έχει θέση σε ένα κράτος δικαίου. Και θα πρέπει η Ρουμανία, η οποία κατά τα τελευταία χρόνια έκανε μεγάλες πρόοδους, να μην οπισθοδρομήσει. Αυτό είναι απαραίτητο, ε, κύριε Επίτροπε, να αναλυθεί η κατάσταση λεπτομερώς και να δοθεί αναφορά ε, στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Γκρίσπεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, δυστυχώς ε, είμαι ε, κρυολογημένη και γι' αυτό θα δώσω τον λόγο στη Σοφίν Βέλτ, θα μου, γιατί δυστυχώς η φωνή μου δεν βγαίνει. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Σήμερα, ε, ναι, εφόσον είστε στον κατάλογο ε, των ομιλητών, δεν μπορώ να δώσω τον λόγο σε άλλο άτομο. Ε, με συγχωρείτε, διότι πρέπει να είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Η Σόφη είναι ήδη στον κατάλογο των ομιλητών, θα μιλήσει αργότερα. Τώρα περνάω στους πράσινους, οι οποίοι δεν είναι εδώ παρόντες. Ο συντονιστής των πρασίνων δεν είναι εδώ. Όχι, όχι, εσείς Είσαστε συντονίστρια, ναι, ναι, ναι. Άλντε πρώτον, θέλετε εσείς συντονιστής της Άλντε να λάβετε τον λόγο για μερικά δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς μερικά στοιχεία πολύ σύντομα για την ομάδα μου και σε σχέση με την κατάσταση στην Ρουμανία θέλαμε η Επιτροπή να διευκρινίσει πράγματι χρησιμοποιώντας ε, στοιχεία αντικειμενικά και δικαιολογημένα όπως υπενθύμησε ο Αντιπρόεδρος στην κατάσταση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης πρώτον και δεύτερον αυτή τη χρήση των ε, μυστικών πρωτοκόλων για τα οποία θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο να έχει εξηγήσει σαφής από την Κομισιό ε, σχετικά με αυτήν ε, την συναλλαγή που φαίνεται να υπάρχει και που φύγει την Ρουμανία μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Σόφινβελτ είναι στον κατάλογο, θα μιλήσει αργότερα. Ο κύριος Ταρικάφρος που είναι συντονιστής των Πρασίνων. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Όχι, όχι. Πρόκειται για τη Ρουμανία και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ε, μιλήστε ίσως ως συντονίστρια, δεν ξέρω. Ναι, ναι, το εκτιμώ αυτό κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω πότε οι πράσινοι άλλαξαν συντονιστές. Αλλά έχω Δύο σημεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ, ερωτήματα που θα ήθελα να θέσω στον Επίτροπο Τίμερμανς. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι είναι δύσκολο να δράστε όταν δεν έχει ακόμα εκδοθεί και κυρωθεί η νομοθεσία. Και θα έχουμε ίσως μια έκθεση την επόμενο μήνα για το επόμενο βήμα. Είδαμε σε προηγούμενες συζητήσεις για την Ουγγαρία και την Πολωνία ότι προτάσεις ήδη αλλάζουν μια κοινωνία και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βρούμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και θα ήθελα να μου πείτε αν σκεφτήκατε την συζήτηση που λαμβάνει ε, χώρα στην Ρουμανία για τον νόμο ε, για ε, τις δημόσιες συναθρήσεις για τους ανθρώπους που μαζεύονται στους δρόμους ε, και φωνάζουν τις ανησυχίες τους. Το δημοψήφισμα επίσης για μια περιοριστική, περιοριστικό ορισμό του οικογενειακού δικαίου. Δημοψήφισμα που θα λάβει χώρα το Σάββατο και την ε, Κυριακή για να αυξηθεί ο αριθμός των ατών συμμετεχόντων στο δημοψήφισμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε επαφή με την κυβέρνηση της Ρουμανίας για αυτό το δημοψήφισμα και ποιο ήταν το μήνυμά σας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Μα δεν μπορείτε ταυτόχρονα να είστε αντιπρόεδρος ε, και ε, συντονίστρια. Τότε φεύγω από αντιπρόεδρος. Φύγετε τότε. Δεν μπορείτε να είστε και τα δύο. Είναι προφανές. Για την ΚΟΕ συντονίστρια για την ΚΟΕ δεν είναι παρούσα. Τώρα περνάμε στην EFDD, Λόρα Φεράρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι, ανησυχούμε ιδιαίτερα για την κατάσταση στη Ρουμανία. Θεωρούμε ότι η αναθεώρηση του ποινικού κώδικα οδηγεί σε παρεμβάσεις στο δικαστικό τομέα και αδυνατίζει, αποδυναμώνει την ε, δικαστική συνεργασία με άλλες χώρες, έτσι ώστε η Ρουμανία να είναι ένας ασφαλής λιμένας για να μπορεί κανείς να προωθεί διάφορες παράνομες δραστηριότητες. Δυστυχώς υπάρχει ε, ατιμορρησία για τους υπεύθυνους πλησίματος ε, χρήματος και επίσης ε, το γεγονός ότι οι υπόδικοι δεν μπορούν να κατέχουν δημόσια αξιώματα. Επίσης γίνεται μία αποποινικοποίηση δυστυχώς της διαφθοράς. Εγώ ήμουνα η συγγήτρια επί του θέματος και είχαμε μιλήσει για την διαφθορά ζητώντας μία επαλήθευση χώρα προς χώρα για ενδεχόμενες παραβιάσεις αυτό αφορά και τη διαφορά Ποιος έχει καταδικαστεί μία φορά δεν μπορεί να, ε, να έχει πρόσβαση σε δημόσιο αξίωμα. Αυτό αφορά και την έκθεση Κοράου που αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η δράση και τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν πολύ καλά αυτό το μηχανισμό και να ρίξουμε φως για το τι συμβαίνει στη Ρουμανία ως προς την τήρηση του κράτους δικαίου. Ο κύριος Ζέστρα από το ΙΕΝΕΦ δεν είναι παρόν. Τώρα, κατάλογος των ομιλητών. για 1,5 λεπτό ανάλογα με το πότε δηλώσατε συμμετοχή. Η κυρία Μακοβέη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα που δεν συζητήθηκε γιατί ανέκυψε χτες και σήμερα. Η ανεξαρτησία του τύπου διατρέχει μεγάλο κίνδυνο. Ο πρόεδρος του ΠΣΕΤΕ, ο ε, Λίβιου Ντράγνε, μίλησε για νομοθετικά μέτρα για την ε, περιστολή των δικαιωμάτων του τύπου. Ήδη γίνονται αιτήσει online κατά αυτής της νομοθετικής ε, πράξης. Πέρα δηλαδή από την ανεξαρτησία του δικαστικού, τώρα έχουμε και το θέμα της ανεξαρτησίας του τύπου, που και αυτή ενοχλεί. Ως προς τη βία ήδη αναφερθήκαμε. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει ε, προσφυγή στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω ποιος έδωσε την εντολή για τα βία αυτά επεισόδια. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Ως προς την αλλαγή του ποινικού δικαίου θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα δηλαδή ο περιορισμός έρευνας μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή, αν μία έρευνα δεν έχει διαλευκανθεί σε ένα χρόνο, τότε σταματάει, γιατί έληξε ο χρόνος. Αυτό αφορά έγκλημα, ε, διασυνοριακό κρίμα, διαφθορά, διασυνοριακές παραβιάσεις. Δεν μπορούν να ερευνηθούν μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό δεν αφορά μόνο τη Ρουμανία. Έχω ακόμα. Έχω 8 λεπτά, λέει η κυρία Μακοβέη. Άρα δεν είναι θέμα της ε, Ρουμανίας αποκλειστικά. Σας διακόπτω γιατί υπερβήκατε το 1,5 λεπτό. Η κυρία Γκραπίνη. 1,5 λεπτό έχετε κυρία Μακοβέη, όχι 8. Γκραπίνη, ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, ξέρω ότι γνωρίζετε την κατάσταση στη Ρουμανία, Έχει, την έχετε επισκεφθεί πολλές ε, φορές. Θα ήθελα να ρωτήσω, απόψε η Επιτροπή της Βενετίας, η Επιτροπή μίλησαν με τα μέλη του ε, συνταγματικού γιατί ελέγχθη δημοσία ότι υπάρχουν απειλές ε, δικαστές και ο Τόνι Γκρέμπλερ καταδικάστηκε πρόσφατα και τώρα είναι ελεύθερος γιατί δεν υπήρξαν αποδεικτικά στοιχεία. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να μου εξηγήσετε είναι γιατί θεωρείτε ε, ότι η Ρουμανία δεν τηρεί το κράτος δικαίου τη στιγμή που μιλάμε για ένα πλαίσιο που ισχύει για το συνταγματικό δικαστήριο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόνι. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, θα έπρεπε να ασχοληθούμε σοβαρά με τη συνθήκη και τα καθήκοντά μας και τις αξίες μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλες τις χώρες μέλη με τον ίδιο τρόπο. Και πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές ανησυχίες όσον αφορά την Ρουμανία. Έχουμε ανθρώπους που διαδηλώνουν στο δρόμο, έχουμε σοβαρές διαμαρτυρίες εκ μέρους των ΜΚΟ ε, έχουμε προβλήματα όσον αφορά το πλουραλισμό των ΜΜΕ στη Ρουμανία και την ελευθερία του τύπου. Έχουμε επίσης προβλήματα όσον αφορά την πάταξη της διαφθοράς. Άρα πιστεύω ότι η κατάσταση είναι αρκετά ξεκάθαρη και επίσης οι ρουμανικές αρχές ε, υπονομεύουν την ε, αξιολόγηση του δικαστικού σώματος. Θα πρέπει λοιπόν όλοι, όλα τα ευρωπαϊκά όργανα και η Επιτροπή να εξεύρει τα ενδεδειγμένα εργαλεία ώστε να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Γιατί ε, όταν ε, θα, η Ρουμανία θα πρέπει να εξαλειφθεί όσον αφορά ε, για παράδειγμα το κράτος ε, δικαίου θα πρέπει ήδη να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ευχαριστώ κύριε πρώτε αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε που παρευρίσκεστε εδώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί παρακολουθείτε εκ του σύνεγγης την κατάσταση στη Ρουμανία και τις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού. Σε όλες τις εκθέσεις ε, CM, CVM, ε, μέσα στο μηχανισμό ε, συνεργασίας και επαλήθευσης, δεν έγινε λόγος για καμία κατάχρηση ή παραβίαση ο μηχανισμός δεν αναφέρθηκε σε τίποτα τέτοιο. Υπήρξαν καταχρήσεις ε, εξαιτίας των ε, ε, κρυφών πρωτοκόλων, αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε ποια αποδεικτικά στοιχεία είναι συναφή και ποια όχι και σε ποια στοιχεία θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση. Νομίζω ότι αν αυτός ο μηχανισμός συνεργασίας και επαλήθευσης δεν είναι αποδοτικός, τότε ας εξαφανιστεί. Αν είναι καλός, ας τον εφαρμόσουμε σε όλα τα κρατη για να δούμε τι συμβαίνει και στα άλλα κράτη-μέλη, όπως λέει ο ΩΣΑ και η Transparency International. Να δούμε ποιοι παραβιάζουν, ποιοι χρηματίζονται και ποιοι όχι. Αλλά παντού αυτά. Η κυρία Ιντβέλτ. Yes, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή τονίζει και πάλι την ε, κατεπίγουσα ανάγκη για έναν ε, μηχανισμό ο οποίος να εξετάζει όλες τις χώρες γιατί αυτό το είδος ε, συζήτηση τελικά καταλήγει με το να στελιτεύουμε ορισμένους, να υπάρχουν αρνήσεις από την άλλη πλευρά, κατηγορίες κλπ. Ε, και δεν υπάρχει καμία λύση. Άρα θα πρέπει η Επιτροπή να κάνει μια πρόταση στην κατεύθυνση αυτή. Όσον αφορά τα συγκεκριμένα προβλήματα, ανησυχώ πολύ για τα προβλήματα που ανέλησε η Επιτροπή, αλλά λείπουν δύο στοιχεία. Η αναφορά στο δημοψήφισμα. Ε, πιστεύω ότι όλα τα προοδευτικά κόμματα θα πρέπει να πούν ε, κατά πόσο είναι υπέρ των ίσων δικαιωμάτων για όλους. Δεύτερον, η διάλυση των ΜΚΟ ε, αφορά και τη μεταφορά της οδηγίας κατά του ξεπλήματος χρήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά των μη κυβερνητικών οργανώσεων η ρουμανική κυβέρνηση, η ίδια ρουμανική κυβέρνηση θα έπρεπε να καλέσει και πάλι την Επιτροπή της Βενετίας προκειμένου να εξετάσει τις μεταρρυθμίσεις έτσι όπως βρίσκεται στο τραπέζι αυτή τη στιγμή πριν τις ε, υιοθετήσει. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να αναστρέψει, να πάρει πίσω τους τα νομοσχέδια που περιορίζουν την ελευθερία των ε, λόγου και, και, ε, κίνησης των μη ε, τέλος, ε, η έκθεση για την ε, διαφορά είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί δείχνει πόσο κατεπίγουσα εδώ είναι η ανάγκη παρέμβασης. Tak, panie przewodniczący, jest mi strasznie przykro, że, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι κρίμα που πάλι συζητούμε για ένα κράτος μέλος και για προβλήματα κράτους δικαίου. Είχαμε την Πολωνία, είχαμε την Ουγγαρία, τώρα έχουμε την Ρουμανία. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση θα ήταν να έχουμε την ίδια προσέγγιση προς όλες τις χώρες που σαφώς υπονομεύουν το κράτος δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάνω έκκληση λοιπόν στους συναδέλφους ε, των σοσιαλιστών και δημοκρατών να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όπως κάνουμε και εμείς στο ΕΛΚΑ, αποφεύγοντας ε, μια κομματική προσέγγιση και να εξετάσουν τα θέματα προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θίγονται αυτά τα συμφέροντα. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αλλαγές εισήχθηκαν στον ποινικό δίκαιο και στον κώδικα ποινικής δικαιονομίας που καθιστά την διασυνοριακή συνεργασία με την Ρουμανία δύσκολη αν ο νέος νόμος για την δικαιοσύνη υπονομεύει την ανεξαρτησία των δικαστών προβλέπεται την ενεργοποίηση του άρθρου 7 και την παραπομπή της Ρουμανίας στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Καρμαρακιούρε. Ναι, Συμφωνούμε όλοι ότι η Ρουμανία είναι μια χώρα πάρα πολύ σημαντική. Σημαντική για την συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι η Ρουμανία έλαβε μέρος στο θέμα σχετικά με τον Σκρίπαλ Ε, πράγμα που δεν έκανε το Βέλγιο ή η Αυστρία. Η Ρουμανία ήταν ε, με το μέρος μας, με το υποστήριξε την ασφάλειά μας και αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μας και η φωνή των συναδέλφων μας σε άλλα κοινοβούλια είναι σημαντική. Ό,τι αφορά τη Ρουμανία είναι σημαντικό. Αλλά έχω μια ειδική ερώτηση για τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαντς. Κατάλαβα καλά ότι κατακρίνατε τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ρουμανίας και ότι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υποστηριχθεί η πολιτική θέση του Προέδρου της Ρουμανικής Δημοκρατίας, λέει η κυρία Λόρα Κέβεση. Και ε, ένα άλλο σχόλιο. Θα περίμενα ο Αντιπρόεδρος να επιβεβαιώσει την ουδετερότητα της Επιτροπής για τέτοια θέματα όπως είναι το οικογενειακό δίκαιο στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ε, βλέπω ότι υπάρχει εδώ πολύ συναισθηματισμό. Σας επανέλθουμε στα σημαντικότερα. Ε, κύριε Επίτροπε, η ερώτησή μου σε σας και ε, μπορεί και που επιβεβαίωσε η Επιτροπή της Βενετίας ποια είναι η σημαντικότερη παραβίαση που θα μπορούσε να οδηγήσει στο να σκεφτούμε ότι η Ρουμανία δεν είναι ένα κράτος όπου τηρούνται οι νόμοι, δεν είναι ένα κράτος δικαίο. Τι πηγές πληροφοριών χρησιμοποιήσατε για να αξιολογήσετε την τρέχουσα κατάσταση ε, στη Ρουμανία. Λέτε ότι επιδεινώνεται η κατάσταση. Μπορείτε να διευκρινίσετε. Επίσης το οικογενειακό δίκαιο είναι κάτι ε, το εθνικό και θα έπρεπε να αποφασίσουν οι πολίτες της Ρουμανίας. Ευχαριστώ. Η ε, Ρουμανία έκανε πολλές πρόοδους στην καταπολέμηση της διαφθοράς και ελπίζουμε ότι αυτό δεν σταματήσει στο μέλλον. Βεβαίως, καλά έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν αρκεί να συγκεντρωνόμαστε σε ιδιαίτερες περιπτώσεις διαφθοράς. Θα έπρεπε να εξετάσει κανείς λεπτομερώς και ενδελεχώς πώς λειτουργεί το κράτος δικαίου και η δικαιοσύνη. Να έχουμε ε, παράνομες αποφάσεις ε, το μετά ε, την ένταξη της χώρας. Μια διαδικασία σταμάτησε και υπήρξε εκεί επανεθνικοποίηση σχετικά με την Ουγγρική Εκκλησία. Ε, το, ε, το, η σχολή ιατρικής επίσης θα έπρεπε να έχουν ένα τμήμα με την μειονοτική Ουγγρική γλώσσα. Για δέκα χρόνια το κράτος επέτρεψε στην, στο Πανεπιστήμιο να παραβιάσει τον νόμο, αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα όπου ε, εφαρμόζεται επιλεκτικά η νομοθεσία, όπως το δικαίωμα μιας δίκαιης δίκης ε, και επίσης ε, τα θέματα της χρησιμοποίησης των συμβόλων της μειονότητας. Όλα αυτά τα θέματα έχουν σχέση με το κράτος δικαίου. Με συγχωρείτε ε, που δεν μπόρεσα να μιλήσω στην δική μου γλώσσα, την Ουγγρική, διότι δεν υπάρχει μετάφραση. Ευχαριστώ. Γκουράνου. Ευχαριστώ πολύ τον Αντιπρόεδρο Μέρμανς για αυτή την παρουσίαση. Ε, γνωρίζουμε πολύ καλά τα γεγονότα της 10ης Αυγούστου και το ρόλο του κράτους. Ήταν ένα τραγικό σύμβαν Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ταπεινώθηκαν από μια κυβέρνηση που δεν μπόρεσε να τηρήσει τα ελάχιστα όρια αξιοπρέπειας. Δεν αντιμετώπισε στο στάτους διαδηλωτές, άσκησε βία η οποία ήταν ανέτεια. Τις επόμενες ημέρες αυτοί οι άνθρωποι ταπεινώθηκαν, ελέγχθη ότι ήταν αρκομανείς, ότι προσπαθούσαν να προωθήσουν ένα πραξικόπημα ή παραστρατιωτικές δραστηριότητες. Η κυρία ε, Πρωθυπουργός, η οποία δεν μιλάει καλά, ούτε καν καλά τη ρουμανική γλώσσα, έκανε τραγικά λάθη. Και η κυβέρνηση ΠΕΣΕΝΤΕ δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να ε, διαλέξουν ε, είτε τη διαφθορά είτε τη βία και τα δύο πάνε πολύ. Έχουμε άλλους ε, δύο ομιλητές δυνάμει του άρθρου 206, Ρενάτα Βέμπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε για την παρουσία σας εδώ. Αναφερθήκατε στα μυστικά πρωτόκολλα και τις ρουμανικές μυστικές υπηρεσίες που αναφέρονταν ότι εναπόκειται στο Κοινοβούλιο να ρυθμίσει το πώς συμπεριφέρονται οι υπηρεσίες πληροφοριών σε μια χώρα. Σωστό. Ωστόσο το πρόβλημα είναι ότι οι υπηρεσίε πληροφοριών το έπρεξαν μέσω μυστικών πρωτοκόλων, τα οποία αποκαλύφθηκαν μόνο του τελευταίους 4 ή 5 μήνε, κάτι που αλλάζει ριζικά το τοπίο. Και για να σα δώσω ορισμένα στοιχεία, ορισμένου αριθμού που σα έδωσα ήδη μέσω μια επιστολή μου. Όλα αυτά τα χρόνια από το 2009, σύμφωνα με μια δήλωση του Νοτάτου Δικαστηρίου, από 30.000 αιτήματα ε, υποκλοπής ε, επικοινωνιών μόνο τρία απορρίφθηκαν. Υπάρχει καμία άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιου είδους ε, ποσοστά. Και άλλο παράδειγμα. τι θα γινόταν εσείς ως Επιτροπή, όποιο ήταν, ή όποιο ήταν το αξίωμά σας ε, είσαστε υπό παρακολούθηση για πολλά χρόνια, 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς να το γνωρίζετε. Πώς θα αισθανόσαστε μετά από τα 8 αυτά χρόνια παρακολούθησης. Ποια θα ήταν η δική σας αντίδραση. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και γιατί προσδέτετε σημασία στην κατάσταση στη Ρουμανία. Ορισμένοι όμως Ρουμάνοι αμαυρώνουν την χώρα τους. Δεν ξέρω αν θα το δεχόσασταν στη δική σας χώρα. Μιλήσατε για την ανεξαρτησία του δικαστικού, της ε, δικαστικής εξουσίας. Είχαμε περίπου 5.000 κρυφά πρωτόκολλα από το ΣΕΡΕΙ και 6 εκατομμύρια ε, Ρουμάνοι είχαν ε, παρακολουθηθεί και τους ε, παρακολουθούσε η Υπηρεσία Ασφαλείας. 2.900 δικαστές και 1.812 εισαγγελείς, δηλαδή 60% του δικαστικού σώματος έχουν ε, ανοίξει την διαδικασία έρευνες. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο ε, τηρείται μία σωστή διαδικασία. Μιλήσατε για τη βία, αλλά το 2008 στις ε, ε, Βρυξέλλες ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία από την αστυνομία στις Βρυξέλλες και στην Ισπανία ακολουθήθηκε η ίδια ε, διαδικασία ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Συνάδελφοι, σας είπα για τρεις ομιλητές δύναμη άρθρου 206 Άρα ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Μποστινάρου, ο τελευταίος ε, ομιλητής. Έχετε το λόγο. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ας μιλήσουμε για γεγονότα και για την ομοθεσία της Ρουμανίας. Οι, οι διαδηλώσεις της 10 Αυγούστου, όπως έχουν περιγραφή αφορούν μια παράνομη σύναξη πολιτών και επιτέθηκαν οι διαδηλωτές και 69 αστυνομικούς και ενός του πήραν και το όπλο. Τι θα γινόταν στην Ολλανδία ή στη Βέλγιο αν γινόταν κάτι αντίστοιχο. Μιλήσατε για την, ε, τον Εθνικό Φορέα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, τον ΤΕΝΑ. Ξέρετε ότι γίνονται έρευνες κατά του ε, δικαστικού στην πόλη Πλοϊέστη, όπου έγινε και παραχάραξη στοιχείων. Και τέλος. Γνωρίζετε ότι ο πρόεδρος της Γερουσίας ε, παρακολουθεί το για 7 χρόνια για λόγους εθνικής ασφαλείας, μέρα νύχτα. Λες και ήταν τρομοκράτης ή σαν να ανήκε σε εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά τα στοιχεία στη συνέχεια απομακρύνθηκαν τι είναι η κατάσταση δικαιοσύνης. Αυτό το κατασταλτικό γεγονός είναι απότοκο της άγνοιας της Επιτροπής επί του θέματος. Δεν μπορείτε να μας μιλάτε για μυστικές υπηρεσίες. Τη στιγμή που οι μυστικές υπηρεσίες καταστρέφουν στοιχεία δεν έπρεπε η Επιτροπή να έχει παρέμβει. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την πειθαρχία σας. Τώρα το έχει λόγο ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Τίμερμας. Start Παρακαλώ, θα κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις για, το που δεν πάνε καλά τα πράγματα κατά την άποψή μου, αλλά συμβαίνει πολύ συχνά, οπότε και την κριτική από την Επιτροπή για ορισμένα νομοσχέδια και προσωρισμένες χώρες μέλη. Αυτοί που θέλουν να υπερασπιστούν αυτό το οποίο συμβαίνει πάντοτε κρύβονται πίσω από την, το έθνος τους ή τους ε, πολίτες. Λέτε αν επικρίνεται το νόμο μου, επικρίνεται τη χώρα μου κλπ. Και τους πολίτες. Όχι, επικρίνουμε συγκεκριμένα κάποιες ε, προτάσεις νομοθετικών αλλαγών που πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν πισοδρόμοι σε σχέση με την, ε, τον αγώνα για την πάταξη της τρομοκρατίας και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κάθε φορά που ασκείται μια κριτική λέγεται όχι, αυτή είναι μια επίθεση κατά των πολιτών. Όχι, πραγματικά είναι κατά την άποψή μου σημείο δυναμίας εάν ε, προβάλλει κανείς αυτό το επιχείρημα. Ε, σημαίνει ότι κανείς δεν έχει άλλα πιο στεναρά επιχειρήματα. Είδαμε τον Πρωθυπουργό, την Πρωθυπουργά να το κάνει στην Ολομέλεια πριν από λίγο καιρό και το ακούμε και πάλι σήμερα. Κάτι το οποίο επίσης δεν ισχύει κατά την άποψή μου είναι να κατηγορούμε άλλους, να λέμε και οι άλλοι το κάνουν αυτό, να επεκαλείται κανείς το τι κάνουν και οι άλλοι. Όμως εμείς αυτή τη στιγμή συζητούμε για τη Ρουμανία. Τρίτον, ε, γιατί έχουμε αυτό το μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου. Γιατί κατά την προσχώρηση της Ρουμανίας το 2007 συμφωνήσαμε ότι για αυτά τα δύο μέλη τα οποία προσεχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε υπήρχαν κάποιες αποκλήσεις όσον αφορά το δικαστικό σύστημα και τον αγώνα κατά της διαφθοράς και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης που θα έπρεπε να διορθούν και δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό για να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό υπάρχει αυτός ο ειδικό μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία πολύ συγκεκριμένα και πιστεύω ότι είναι το πιο ενδεδειγμένο εργαλείο ώστε να βοηθεί η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Εμεί μιλάμε για τη Ρουμανία να, ε, να εξασφαλίσουμε ε, οι χώρες αυτές να φτάσουν σε ένα σημείο που ε, το δικοστικό σώμα να είναι αρκετά ισχυρό, όπου η πάταξη τη έχει φτάσει σε ένα μη αναστρέψιμο σημείο κλπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξαφανιστεί εντελώ, αλλά θα υπάρχουν τα, οι μηχανισμοί που μπορούν να επιληφθούν αυτών των θεμάτων. Και τα λέω γιατί, όπως θα ακούσατε ε, από τον κύριο Γιούγκερ, η ε, Επιτροπή ψάχνει ένα μηχανισμό για να ρυθμίσει τα ζητήματα κράτος δικαίου σε όλες τις χώρες μέλη. Αυτό είναι που κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε αυτό το ειδικό μηχανισμό το οποίο δημιουργήθηκε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες ε, στην περίπτωση αυτής της χώρας. Και θα πρέπει να σας πω, αυτό δεν είναι τίποτα καινοφανές, είναι κάτι το οποίο γράψαμε και στην παρεμιζάνη έκθεση το περασμένο Νοέμβριο. Ε, ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια πιστοδρόμηση και αυτό είναι πηγή μεγάλης ανησυχίας. Ε, και δεν θα ήθελα να παραλάβω τα είπα. Νομίζω ότι ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Δεν το λέει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λέει η Επιτροπή της Βενετία. Δεν το λέμε εμεί επειδή έτσι μα κατέβηκε. Και παρακαλώ, ας μπούμε ε, σε ένα διάλογο σχέση με αυτά τα πολύ συγκεκριμένα θέματα. Ας μην αποκλίνουμε, ε, γύρουμε ε, απαιτήσει χειρισμού κλπ. και, νομίζω ότι αυτό θέλει να κάνει η ρωμανική κυβέρνηση. να καθίσει να συζητήσει μαζί μας για την εξέβρεση ενδεχόμενων λύσεων. Το ζήτημα των μυστικών πρωτοκόλων τώρα. Ε, δεν καταλαβαίνω πώς ε, θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το θέμα των μυστικών πρωτοκόλων, τα οποία όλα ε, δημοσιοποιήθηκαν ως πρόσχημα για να δικαιολογήσετε την ε, μεταρρύθμιση της νομοθεσίας η οποία θα περιορίσει, θα υπονομεύσει τον αγώνα κατά της διαφθοράς. Αυτή τη σύνδεση κάνετε. Γιατί την κάνετε. Ωραία, ας το συζητήσουμε ε, και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μία λύση για το θέμα αυτό. Μην επικαλείστε άλλα πράγματα. Τώρα, για τις διαδηλώσεις. Έχουν γίνει έρευνες και ας δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των ερευνών αυτών. Ε, όλοι είδαμε τις εικόνες και όλοι είδαμε επίσης, ακούσαμε τις μαρτυρίες των πολιτών μετά. Δεν ήταν άνθρωποι που θα μπορούσαμε να σχέσουμε ότι είναι χούλιγκαν ή κάποιοι που διαταράσουν τη δημόσια τάξη. Ήταν κάποιοι που διαδήλωναν ειρηνικά. Αλλά, όπως σας είπα, περιμένουμε τα πορίσματα των ερευνών. Τώρα, η οδηγία για το κατά του ξεπλήματος. Ε, η Επιτροπή ε, την Ρουμανία στο δικαστήριο. Τι πληροφορίες έχουμε σε σχέση με τις σοβαρές παραβιάσεις. Νομίζω ότι αναφέρθηκα σε αυτό στην εισαγωγή μου και θα συνεχίσουμε αυτό το διάλογο ε, προετοιμάζουμε εξάλλου τη νέα έκθεση του Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελέγχου. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτό αναφέρεται στο θέμα της ε, οργάνωσης δικαιοσύνης, την ε, διαδικασία απόλυψης του επικεφαλής ε, ε, της υπηρεσίας πάταξης διαφθοράς κλπ. Εγώ είπα ότι ο πρόεδρος της Ρουμανίας ε, δεν ήθελε αυτή την απόλυση, αλλά παρόλα αυτά αυτή ήταν απόφαση του δικαστηρίου. Εγώ δεν επέκρινα κατά κανένα τρόπο την απόφαση του δικαστηρίου. Και όπως σας είπα, ο ποινικό ε, δικονομικός κώδικας ε, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο θα έπρεπε να συζητήσουμε. Και ε, το είπα στην κυρία Μακοβέη, είπατε, ε, στον κύριο Τράκναρ σε σχέση με τα όσα είπε για την ανεξαρτησία των ΜΜΕ. Εάν θα έπρεπε να αντιδρούμε σε οτιδήποτε λένε οι πολιτικοί, ας δούμε καλύτερα κατά πόσο υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση και κατά πόσο υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα λόγο να ανοίξω ένα θέμα για την ανεξαρτησία των ΜΜΕ στη Ρουμανία. Θα ήθελα να περιοριστώ στα ζητήματα τα οποία ήδη έχω αναφέρω. Τώρα, όσον αφορά το δημοψήφισμα για τον οικογενειακό νόμο, για την οικογενειακή νομοθεσία, εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Η, το οικογενειακό δίκαιο αποτελεί η αρμοδιότητα των χωρών μελών δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος σε αυτή την αίθουσα ο οποίος να γύρει κάποιες αμφιβολίες εδώ. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση γενική φύσης που δεν αφορά δηλαδή μόνο τη Ρουμανία, αλλά γενικώ αυτή την επιτροπή. Εγώ πιστεύω πολύ στις οικογενικές αξίες, είμαι ε, σύζυγος πατέρας τεσσάρων παιδιών κλπ. Αλλά δεν θέλω να χρησιμοποιηθεί χρησιμοποιηθούν οι οικογενειακές αξίες σαν ένα όπλο προκειμένου να δικαιολογηθεί η ομοφοβία ή, διάφορες, ε, ή για να πολεμηθούν άλλες ε, μορφές πέραν της ε, γνωστής, του γνωστού σχήματος πυρηνική οικογένεια. Δεν θέλω να επισέλθω στο δικαίωμα της κάθε χώρας προκειμένου να έχει τη δική της νομοθεσία και για παράδειγμα να θεσπίσει ένα νόμο υπέρ ε, του γάμου ε, ομοφιλοφίλων. Εγώ είμαι υπέρ ε, αυτού του μια τέτοια δυνατότητα. Και το δικό μου κοινοβούλιο άλλωστε είναι από τα πρώτα που επέτρεψε τέτοιου είδου ε, σχέσεις. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι αναπόκειται στην κάθε χώρα μέλος να αποφασίσει και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ότι θα πρέπει κάτι τέτοιο να χρησιμοποιείται σαν εργαλείο προκειμένου να ε, ρίχνουμε λάδι στη φωτιά κατά σεξουαλικών ε, μειονοτήτων ή προκειμένου να πάμε τις ε, γυναίκες σε μεσονικές ε, καταστάσεις, κάτι που συμβαίνει σε πολλά μέρη του κόσμου. Το ξαναλέω, όσον αφορά τα θέματα αυτά, σέβομαι πλήρως τα όσα πράττουν οι χώρες σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η, η ισότητα η οποία ε, δράστες στις ευρωπαϊκές συνθήκες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών και να συμπεριλαμβάνει και τις σεξουαλικές προτιμήσεις ε, των πολιτών. Ε, Βεβαίω θα γίνει μια σχετική συζήτηση στην Ολομέλη. Εγώ θα έχω και μια άλλη συζήτηση με την Ρουμάνα Πρωθυπουργό. Ε, μέχρι στιγμής τα μέλη ε, της ρουμανικής κυβέρνησης είπαν ότι ε, θέλουν να συνεχίσουν ένα σοβαρό διάλογο, επικοδομητικό διάλογο με εμάς, παρόλα αυτά δεν υπήρξαν αυτά βήματα. Κατά την άποψή μου και υπό την ιδιότητά μου ως ε, πολιτικού και διπλωμάτη, η Η ίαση της Ευρώπης είναι το πιο καθοριστικό στοιχείο ε, και δεν θα πρέπει να αποκλίνουμε από, τα βασικά, από τις βασικές αρχές ε, που μας έκαναν να ενωθούμε. Και μια τέτοια βασική αρχή είναι το κράτος δικαίου, το οποίο θα πρέπει να κινητοποιηθεί, ε, να ενεργοποιηθεί σε όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, η πάταξη της διαφθοράς είναι ουσιώδους σημασίες προκειμένου να κατοχυρωθούν οι ευρωπαϊκές αξίες. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, για την ε, συζήτηση. Δεν έχουμε τίποτα στα διάφορα. Τέλος της συζήτησης. I've given you answers,